21 η Μαΐου του 2011. Η υπογραφή πράξεων υπό την ε, συνήθη ε, νομική διαδικασία. Πρόκειται για την ε, συνήθι νομική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 74 του κανονισμού. Οι τίτλοι αυτών των νομοθετικών πράξεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά αυτής της συνόδου περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως τροποποιήσεις στην ημερησία διάταξη. Μονάχα ένα αίτημα για την Δευτέρα, δηλαδή για σήμερα. την 1η Ιουνίου η διάσκεψη των Προέδρων επιβεβαίωσε το πρόγραμμα το οποίο έχετε ε, στον φάκελό σας και μπροστά σας. Η ομάδα ε, των φιλελεύθερων δημοκρατών ζήτησε η διαδικασία επιλογής για το διοικητή του Διεθνούς Μεσονοτικού Ταμείου και την εξωτερική ε, εκπροσώπηση του ευρώ να λάβει χώρα αμέσως μετά την έκθεση του κυρίου Λάινεν σχετικά με τους ευρωπαϊκούς περιβαλλοντικούς οικονομικούς λογαριασμούς. Ε, η κυρία Κούλα θα μας ε, παρουσιάσει το αίτημα αυτό, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για ένα αίτημα ε, ε, απλώς καλών τρόπων και ευγενίας έτσι ώστε να επιτρέψουμε στον κύριο Όλι Ρεν να ασχοληθεί με το θέμα των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικονομικών λογαριασμών και αμέσως μετά με το θέμα του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου. Νομίζω ότι είναι καλό, ε, είναι θέμα ευγενίας προς τον Επίτροπο ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θέλει κάποιος να μιλήσει υπέρ του αιτήματος αυτού. Φαίνεται ότι δεν είναι απαραίτητο, δεν υπάρχει λόγος. Κάποιος ο οποίος θέλει να εκφραστεί κατά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ φρονώ ότι το αίτημα αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό διότι δεν ε, θεωρώ ότι υπάρχουν λόγοι να μην δεχτούμε το αίτημα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιο που θέλει να εκφραστεί πλέον κατά τη προτάσεω αυτή. Κάποιο που θέλει να εκφραστεί λοιπόν κατά τη προτάσεω. φαίνεται πως συμφωνούν όλοι. Ποιο είναι υπέρ του αιτήματο της κυρίας Κούλα. Ευχαριστώ, κατά. Αποχές Εγκρίνεται λοιπόν αυτή η τροποποίηση της ημερησίας διατάξεως. Επομένως η διαδικασία επιλογής του νέου διοικητή του ε, ε Διεθνούς Προσδικού Ταμείου ε, και της εξωτερικής ε, προσέγγισης του ευρώ θα λάβει χώρα αμέσως μετά τη συζήτηση της έκθεσης Λάινεν Ευρωπαϊκή Περιβαλλοντοοικονομική Λογαριασμή. Μία μικρή τροποποίηση λοιπόν στη μέση διάταξη μετά από την οποία μπορούμε να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, σύμφωνα με τη μερίσια διάταξη λοιπόν, έχουμε το πρώτο σημείο μας, αφορά δήλωση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, λόγω της επαιτίου των μαζικών εκτοπίσεων του 1941 στα κράτη της Βαλτικής. Μετά από την δήλωση θα ακολουθήσει σύντομος γύρος ομιλητών από τις πολιτικές ομάδες οι οποίες ε, θα μιλήσουν για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε.